Meine Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε αυτήν ε, εδώ την απογευματινή συνεδρίαση, την ε, ε, έκτακτη συνεδρίαση, η οποία τελειώνει στις 9.30 γιατί σήμερα είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο καλοκαιρινό θα έλεγα βραδάκι ε, είναι κανείς που διαφωνεί με την ημερήσια διάταξη. Όχι, δεν έχει και ο πρόεδρος κάτι να πει. Θεωρεί κάποιος ότι υπάρχει λάθος στα πρακτικά, γιατί έχουν ιστορική αξία τα πρακτικά. Τα πρακτικά του Οκτωβρίου, της 19ης Οκτωβρίου. Ich, ε, η επικεφαλής της γραμματέας ε, θα μπορούσε να έχει κάτι πιο κοντά στο μέλλον, κάτι πιο κοντά. Επίσης έχουμε και τα, ε, τα πρακτικά της 22 ε, Σεπτεμβρίου. Αν περιμένουμε άλλους τρεις μήνες θα είχαμε την ετήσια επέτειο. Πάμε τώρα λοιπόν στην έκθεση μία νέα ε, στρατηγική καινοτόμα και, για το μέλλον ε, του εμπορίου και των επενδύσεων. Με προσανατολισμό στο μέλλον η στρατηγική αυτή. Από τον ε, εισηγητή υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Πάμε λοιπόν απευθείας ε, στην ψηφοφορία. Ε, συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 14 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ όλου αυτού του έργου, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. «56 ψήφισαν, 46 υπέρ, 3 κατά, με 7 αποχές εγκρίνεται». Συγχαρητήρια. Ε, πέτυχε ο εισηγητής να μας φέρει πιο κατά προς το τέλος. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα στάνταρ, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Η συγγήτρια, η κυρία Κβίστου Τρόβολ, είναι εδώ. Δεν είναι εδώ για αυτονόητους λόγους. Έχασε τον άντρα της τις τελευταίες μέρες. Πέθανε ο άντρας της. Αν δεν το ξέρετε. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται.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 Συμβαστική α, η τρο, ε, τροπολογία 56. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγώ είμαι κατά. με παραλίγο να μην απορριφθεί, αλλά απορρίφθηκε. Φτάνουμε στη συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 57. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. 57. Τροπολογία 57. Πέρα της ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται. Και 20 αποχές. Η 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 8 σε δύο τμήματα υπέρ για το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία 44 ψήφοι υπέρ. 9 κατά. Σάρλς, υπέρ ή κατά. Αποχή. Συγχαρητήρια. Στην εισηγήτρια που δεν είναι παρούσα. Ερχόμαστε τώρα Εντάξει, με τις ψηφοφορίες. Ωραία. Ερχόμαστε τώρα στην κοινή συζήτηση για το Τουρκμενιστάν. Τρεις είναι οι εκθέσεις. Στην αρχή έχουμε την κυρία Μανέσκου ως εισηγήτρη. you? Thank you, Chair. Yeah. Ευχαριστώ, εδώ είμαι. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα επίμαχο. Και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια θετικότερη προσέγγιση, έχοντας επίσης κατά νου το γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας συζητείται από το 1998. Έχει περάσει πολύ καιρό, ίσως ε, φέτο να την ολοκληρώσουμε και με την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ σχεδόν όλε οι χώρε την έχουν κυρώσει. Το κείμενο που προτείνω είναι ένα συνοδευτικό ψήφισμα με αυτή την ε, συμφωνία Τερκής σχέσης και συνεργασίας. Ε, δεν είναι ιδιαίτερα μακροσκελές ε, το κείμενο, γιατί είχαμε περιορισμό λόγω της διαδικασίας, αλλά όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συνάδελφοι θα καταθέσουν τις τροπολογίες. Νομίζω ότι αυτό το ψήφισμα έχει μεγάλη σημασία, γιατί η επικύρωση τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο για το Κοινοβούλιο, αλλά και στη σχέση με την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Νομίζω ότι εμεί ω Κοινοβουλίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία στο Τουρκμενιστάν, ζητώντα λεπτομερεί εκθέσει και δεδομένα. για αυτό το φάκελο. Είχα πολλές ε, συνεδριάσεις, συνεργάστηκα στενά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ανησυχούν ιδιαίτερα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Με βοήθησαν ε, πάρα πολύ, καθώς παρήχαν χρήσιμες πληροφορίες και έγγραφα. Επίσης, έχω εργαστεί πολύ καλά με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τον ειδικό αντιταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία, τον κύριο Μπουριάν. Νομίζω ότι η όλη εμπειρία ήταν πολύ σημαντική, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να έχουμε μία σαφή και ξεκάθαρη εικόνα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή τη Συμφωνία Εντερικής Σχέσης και Συνεργασίας, έχω συστήσει στο κείμενο να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπω να έχουμε πέντε κυρίες πτυχές. Και πολύ σύντομα θα θέλω να τις υπογραμμίσω. Η πιο σημαντική είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που ήδη διευθυντήθηκε από το Τουρκμενιστάν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει διατάξεις για το μηχανισμό παρακολούθησης και ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα είναι νομικά υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, έτσι όπως ε, αναφέρεται στο εθνικό σχέδιο. Επίσης, θεωρήσα ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Τουρκμενιστάν. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια γενική στρατηγική. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τη νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία, η οποία συγκεκριμένα αναφέρει ότι κάθε στρατηγική θα πρέπει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό είναι κάτι καινούργιο και θα βοηθήσει και το Τουρκμενιστάν. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη χώρα που έχει συγκεκριμένα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στην εκπαίδευση. Στα σχέδια εκπαίδευσης προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το έδαφος για καλή συνεργασία με το Τουρκμενιστάν. Θα μάθουμε και από τα λάθη μας σε ό,τι αφορά άλλες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, παραδείγματος χάρη. Και αν αντλήσουμε κάποια διδάγματα, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη μας πιθανότατα. Είναι καλό που έχουμε αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μεν, αλλά είναι κάτι που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν δε. Επομένως, χρειαζόμαστε το δικό μας μέσο για να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτού και η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας θα μας προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης αυτής της εφαρμογής. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα θετικό βήμα, το αναγνωρίζουμε, δηλαδή το ότι έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Είναι κάτι που γίνεται από την κυβέρνηση. Δεν είναι όμως δεσμευτικό, ούτε έχει όρους ε, πολλαπλή συμμόρφωσης. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε πολλαπλή συμμόρφωση, και αν θέλουμε να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει μια μεταρρύθμιση στον τομέα των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, χρειαζόμαστε ένα μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. φυσικά η PCA, η Συμφωνία Ατρικής και Συνεργασίας, μπορεί να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Θέλω να αναφερθώ και στο στρατηγικό ρόλο του Τουρκμενιστάν ως ουδέτερο κράτος σε ό,τι αφορά την περιφερειακή σταθερότητα. Δεν θα πρέπει αυτό να το παραμελήσουμε. Είναι πολύ σημαντική πτυχή και το ότι το Τουρκμενιστάν είναι μέλος σε διάφορους οργανισμούς, συμβάλλει στην αναγνώριση της διεθνής του προσπάθειας ε, για παγκόσμια ανάπτυξη. Θα, θα επιλέξει τους συμμάχους του σύντομα το Τουρκμενιστάν. Είναι λοιπόν πολύ πιο βολικό για μια χώρα που δεν θέλει να κάνει μεγάλες αλλαγές, να επιλέξει τους συμμάχους που δεν ε, θέτουν προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να τους έχουμε με το μέρος μας και να κατανοήσουμε ότι τώρα είναι το παράθυρο ευκαιρίας της Ευρώπης για να δεσμευτούμε και εμείς ότι είμαστε τέρος για το Τουρκμενιστάν. Με όλες τις προϋποθέσεις φυσικά όλους τους όρους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας και τα αιτήματά μας ως εταίρο. Το τρίτο σημείο. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών στο Τουρκμενιστάν και που έχουν τώρα την ευκαιρία να λάβουν τη βοήθειά μας για τις δραστηριότητές τους, είναι και αυτή μια πτυχή που δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε. Υπάρχουν ε, πολλές ενώσεις που έχουν εγγραφεί το 2014 και το 2015. Η δραστηριότητά τους αυτή τη στιγμή περιορίζεται σε κάποιους τομείς, όπως ε, του να υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, ε, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, παροχή νομικής βοήθειας για θέματα εμπορίας ανθρώπων και οικοδόμηση δυνατοτήτων για τη οργανώσει κοινωνία των πολιτών. Έτσι λοιπόν, είναι καλό να σκεφτούμε ότι μέσω τη PCA, μέσω του μέσου που προτείνουμε προ επικύρωση, να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτέ τι οργανώσει και θα συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε και να τις βοηθήσουμε να μεγενθηθούν. Και δεν μιλώ μόνο για αυτές τις οργανώσεις, αλλά αυτό είναι μια αρχή. μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερε οργανώσει κοινωνικών πολιτών και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορούν να υπάρχουν στη χώρα. Ένα άλλο ζήτημα είναι τα σημερινά προγράμματα δημιουργού συνεργασία στο Τουρκμενιστάν. Αυτή τη στιγμή η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τρέχει ορισμένα προγράμματα με το Τουρκμενιστάν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και μέσω της PCA, της Συμφωνίας Ιταρικής Σχέσης και Συνεργασίας, μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας και να διευρύνουμε την επιρροή μας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η οικονόμηση δυνατοτήτων, στο διοικητικό τομέα, που σε μια χώρα όπως το Τουρκμενιστάν νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία για μας, ως εταίρους, και τη συνιστόσα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, οργανώσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων και υπηρεσιών. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα project είναι ουσιαστικά για να τα συζητήσουμε και να εντοπίσουμε λύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πιστεύω ότι η επικύρωση της συμφωνίας θα ενδυναμώσει τη συνεργασία επί αυτών των έργων. Ένα ακόμη σημείο έχει να κάνει με το νέο σχέδιο συντάγματος. Προτάθηκε ήδη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό το σχέδιο συντάγματος θα ήταν καλό να είχε λάβει μια γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ίσως αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Και εγώ θα καταθέσω προσωπικά μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτή η επικύρωση αναβλήθηκε ήδη για πάρα πολύ καιρό. Και αν πράγματι θέλουμε να δεσμευτούμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε το λαό του Τουρκμενιστάν και να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, πρέπει να είμαστε παρόντες. Αν δεν είμαστε παρόντες, αν μόνο θέτουμε τις προϋποθέσεις και περιμένουμε παόριστον να τις υλοποιήσει η κυβέρνηση, τότε δεν είμαστε ρεαλιστές. Και τελικά δεν θέλουμε να βοηθήσουμε το λαό. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε το λαό, θα πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες με το μέσο που παρέχει η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Έχω ζητήσει, όπως θα δείτε, στο σχέδιο ψηφίσματος να έχουμε και μία πλήρη αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αυξήσει το επίπεδο της δικής μας αντιπροσώπευσης στο Τουρκμενιστάν και θα θεωρηθεί ως η δική μας δέσμευση στο να υποστηρίξουμε το Τουρκμενιστάν ως εταίρο στην περιοχή. Θα συνεχίσω να εργάζομαι στενά με τους συναδέλφους, τους και εισηγητές και καλωσορίζω τις τροπολογίες και τα σχολιά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Προτείνω τώρα να συζητήσουμε τα σημεία 6, 7 και 8 σε κοινή συζήτηση και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπουριάν, ειδικό ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να έχω ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές για την επικύρωση της συμφωνίας, τερικής σχέσης και συμφωνίας με το Τουρκμενιστάν. Θα συζητήσουμε επίσης τις εξελίξεις στη χώρα. Η συγγήτρια κυρία Μανέσκου είπε ήδη πολλά σημαντικά πράγματα, οπότε εγώ θα είμαι σύντομος. Θα σας δώσω και τις προσωπικές μου εμπειρίες από την επισκέψή μου στο Τουρκμενιστάν. Τρεις φορές το έχω επισκεφθεί από τότε που ορίστηκα ως ειδικό ε, εκπρόσωπος ε, πέρυσι και έχουμε ξεκινήσει έναν εντατικό ανοιχτό διάλογο για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με τους εκπροσώπους της χώρας. Ε, να σας πω ότι προσφάτως Κατέγραψα το μεγάλο ενδιαφέρον των αρχών του Τουρκμενιστάν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στους τομείς όπου κατά το παρελθόν η ηγεσία του Τουρκμενιστάν ε, δεν ήθελε, ήταν απρόθυμη να έχει κάποια συνεργασία. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα θετικό δείγμα ε, μια, ενός προοδευτικού ανοίγματο ε, της κοινωνίας. Υπήρξαν και μεταρρυθμίσεις στο, στη δεύτερη θητεία του Προέδρου. Η χώρα αυτή, όπως γνωρίζετε, από τη στιγμή που ε, έγινε μια ανεξάρτητη χώρα είχε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, πολλά προβλήματα. Η πρόοδος ε, των μεταρρυθμίσεων ε, και των αλλαγών, πρέπει να πω ότι εξακολουθεί να είναι βραδία και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο πρόεδρος Μπέντι Μουχάμιντοφ ενέκρινε σταδιακά μέτρα που ανέτρεψαν τα πιο καταστροφικά αποτελέσματα των αποφάσεων και της πολιτικής των προκατόχων του. Και στόχος του Προέδρου είναι να μπει στο διεθνές προσκήνιο για το Τουρκμενιστάν και να διαδραματίσει όλο και περισσότερο ενεργό ρόλο. Εκεί Παραδείγματο χάρη όπως ε, στην περίπτωση των έργων υποδομή στο Αφγανιστάν, συνδέσεις, ηλεκτροδότηση, μεταφορέ για να επηρεάσει την κατάσταση στη χώρα. Αυτή είναι η πρόθεση του Πρόεδρου. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή στη χώρα. Έχει εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις περιορισμένες όμως, αλλά Τουρκμένοι φύνοντες πλέον πρέπει να διαφοροποιήσουν την οικονομία λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ξέρουμε ότι υπάρχει πλήρης εξάρτηση από τι εξαγωγέ φυσικού αερίου. Το είπε και η συγγήτρια κυρία Μανέσκου ότι εδώ πλέον διανοίγονται νέοι ορίζοντε για εμάς για να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τουρκμενιστάν τη θεωρεί αξιόπιστο εταίρο για τι προσπάθειε εξυγχρονισμού τη χώρα. Βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματο, ελκυστικότητα για τι επιχειρήσει, επενδύσει, νέε τεχνολογίε. Και τέλο, το Τουρκμενιστάν και άλλες χώρες της περιοχής θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα παράγοντα εξισορρόπησης ε, για την Κεντρική Ασία. Έχουμε την παρουσία της Ρωσίας από πλευράς ασφάλειας και την παρουσία της Κίνας από πλευράς οικονομικής δύναμης και μπορεί να παίξει το ρόλο του εξισορροπητή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο ενεργό ρόλο στη χώρα, να στηρίξει τον εξυγχρονισμό και την αλλαγή βάση των οικουμενικά αποδεκτών αξιών και αρχών. Στις επισκέψεις μου, στο Τουρκουμενιστάν απέδωσα πολύ προσοχή στα ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στην πλευρά ε, και κυρίως στον Υφυπουργό ε, στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση ε, ήμουν πολύ ανοιχτό. Ήταν και η ίδια ανοιχτή ο Σω. συζητούσαμε αυτά τα θέματα, δεν συμφωνούσαμε και σε όλα πάντως ε, έδειξαν ε, ότι είναι πιο πρόθυμοι και διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν ε, σοβαρά και πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πάντα στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική χρονική στιγμή γιατί άπαξ και αναγνωρίσεις ότι έχεις πρόβλημα μπορούν οι εταίρες να σε βοηθήσουν να βρεις και τις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι δεν αρνούνται πλέον ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και αυτό φέρεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπε και η κυρία Μανέσκου. Το κείμενο αυτό βασίζεται στις συστάσεις ε, της Οικουμενικής Περιοδικής ε, Εξέτασης. Εμείς τονίσαμε από πλευράς μας την σημασία Δημιουργία ενό ε, μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου ε, και επίσης θεωρούμε ότι και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ε, θα πρέπει να συμμετέχει στη συνταγματική μεταρρύθμιση. Ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες η Αρμόδια Επιτροπή. Θετική ήταν και η ανταπόκριση ως προς αυτή την πρόταση, άρα νομίζω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για πιο στενή συνεργασία. Δεν θέλω βέβαια να είμαι υπεραισιόδοξο, ε, ούτε να, να υπερτιμήσω τις εξελίξεις. Στο σχέδιο έκθεσης αναφέρονται διάφορα ζητήματα ε, στη έκθεση του Κοινοβουλίου για την στρατηγική για την Κεντρική Ασία, ότι δηλαδή θα πρέπει την ε, όλη διαδικασία να την ε, μετρήσουμε με γνώμονα τα πρακτικά αποτελέσματα και να μην μένουμε στις δηλώσεις, αλλά νομίζω ότι τα πρώτα βήματα είναι θετικά. Και σίγουρα και η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία, όπω υπόθηκε, θα μα δώσει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και μια νομική βάση για μια συνεχιζόμενη ανταλλαγή απόψεων και ελπίδα με το Τουρκμενιστάν. Επίσης πιστεύω και συμφωνώ και με αυτό που είπε η κυρία Μανέσκο ότι δηλαδή η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ε, ανταμοιβή ή βραβείο προς το Τουρκμενιστάν απλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πιο στενής συνεργασίας που θέλει να προωθεί τις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων θα είναι και ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς έχουν δεσμευτεί και δύο πλευρέ. Έχουν συγκεκριμένε δεσμεύσει αναλάβει. Υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξει Τέλος, η συμφωνία αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να ε, δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ενισχυμένου διαλόγου σε όλα τα θέματα και για τη συνεργασία μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στη δημιουργία μια κοινοβουλευτική επιτροπή για τη συνεργασία. Όταν λοιπόν αρχίσει να ισχύει αυτή η συμφωνία και εδώ ολοκληρώνω μια ε, κοινή, ε, επιτροπή τη κοινής επιτροπής, ε, της επιτροπής ετησίω, ε, μέχρι στιγμή δεν μπορούσαμε να εργαστούμε πιο συστηματικά. Τώρα νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πιο στενέ επαφέ και με ε, άλλους ε, βέβαια φορεί, ε, όπως είναι και η κοινωνία των πολιτών, το είπα και στην πρόσφατη συνάντηση, υπάρχει άνοιγμα και περιμένει και η άλλη πλευρά αυτή την πιο στενή συνεργασία. Αυτά ε, ήθελα να σας αναφέρω ε, επιπροσθέτω στον όσον ανέφερε ήδη η συγγήτρια κυρία Μανέσκου και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας ε, να ακούσω τα σχόλιά σας και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούριαν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση πρώτος ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μανέσκου για την έκθεσή της ότι αφορά τη σύναψη τερικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν. Πράγματι, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να βελτιώσει, να αναβαθμίσει στρατηγική της για τη συνεργασία με την ε, Κεντρική Ασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε και στα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Έχουμε και την έκθεση για την αναθεώρηση και υλοποίηση της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Ασίας. Θα την ψηφίσουμε αυτή την εβδομάδα. Όπως υπόθηκε και από τη συνάδελφη και από τον κύριο Μπουριάν, έχουμε το θέμα ε, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν, που ε, δεν είναι ακόμα στην ιδεατή κατάσταση, στο ιδεατό ε, επίπεδο, ε, οργάνωση εκλογών και πολλά άλλα πόρα που έχουν των ε, προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να ενισχύσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και θα πρέπει να επιλέξουμε τη δράση και αυτήν την αδράνεια για αυτό το σκοπό. Συμφωνώ λοιπόν στα μια, μάλλον υπάρχει μια αντιπροσωπεία ε, της ε, Ένωσης ε, για να μας βοηθά να καταλαβαίνουμε την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν και να προωθεί τα θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας, Συμβούλιο, Επιτροπή Συνεργασίας, όλα αυτά προβλέπονται από αυτή τη συμφωνία τέρικης σχέση και συνεργασία και θα ε, βελτιώσουν, θα βελτιώσουν τη δουλειά μας εκεί. Επίσης, ε, μηχανισμός εποπτείας, παρακολούθησης, Ελπίζω να έχει συμμετοχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μα δώσει και αυτό ο μηχανισμό τη δυνατότητα να παρακολουθούμε εκ του σύνοικη τι εξελίξει ε, στο Τουρκμενιστάν, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με το άρθρο 2.2 Τη συμφωνία. Ξέρετε ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στο Κοινοβούλιο σε αυτό το άρθρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Μανέσκου, τη συνάδελφό μας και τον κύριο Μποριάν. Εγώ θα είμαι λίγο πιο ανοιχτό μεν, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με αυτή την έκθεση που πρέπει να απαντηθούν κατερχούν Καταρχάς, μπορεί να, να υπάρχει μια ηθελημένη απόφαση να καθυστερήσουμε την συμφωνία με το Τουρκμενιστάνος τώρα και αν θέλουμε ε, να την προχωρήσουμε τώρα, ε, θα πρέπει να δούμε τι είναι καλύτερο σήμερα από ότι ήταν στο παρελθόν που καθυστερούσαμε την ε, έγκριση. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι κανείς εδώ σοβαρά θεωρεί ότι μπορούμε να πεμπλακούμε από χώρες όπως το Τουρκμενιστάν. Υπάρχει όμως ένα μνημόνιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκμενιστάν και πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τι μπορούμε μαζί να επιτύχουμε μέσα από τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας δρώντας ε, μαζί βάσει του μνημονίου. Τρίτον, όταν μιλάει η κυρία Μανέσκου για τα λάθη στην Ανατολική γειτονία, μάλλον ε, λίγο υποβαθμίζει το γεγονός ε, εσκεμένα, όμως πρέπει να προσέχουμε. Σωστά λέει, ότι υπάρχουν παραλληλισμοί με άλλες χώρες, όμως καλό θα ήταν να αποφεύγουμε να λέμε πράγματα για το Τουρκμενιστάν που θα μας ε, ε, έκαναν να το σχετίσουμε με άλλες χώρες. Αυτό ίσως καλό θα ήταν να το κάνουμε μόνο σε ιδιωτικές συζητήσεις, όχι δημοσίως. Υπάρχει πάντοτε ε, υποψία εξαιτίας της ε, συνεργασίας της ενεργειακής που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Τουρκμενιστάν υπάρχει υποψία ότι θα κάνουμε τα στραβά μάτια για τα ανθρωπίνα δικαιώματα και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην ημερήσια ε, διάταξη να δούμε το μεγάλο αριθμό των εξαφανίσεων, τους πολιτικούς κρατούμενους, τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, τις διάφορες διαδικασίες που έχουν μπλοκαριστεί τα, τα τις ανεξάρτητες ε, διαδικασίες για τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, την καταστροφή του υλικού της δορυφορικής τηλεόρασης. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν στα αρχεία και αυτό ε, πρέπει να το καταγράψουμε για να μην αποσιωπηθούν, οι επικρίσεις που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Όσον αφορά τώρα στην κοινωνία των πολιτών, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την καταγραφή των ανεξάρτητων ΜΚΟ και την υποστήριξή τους από εμά, θα υπάρχει πραγματικά αλλαγή. Και αν αυτό το κάνουμε και συλλογικά, ε, η συγκέντρωση θα έχει την υποστήριξή μου. Τέλος, για την αποστολή, την αντιπροσωπεία. Οι φίλοι μου στο ΕΛΚ πολύ συχνά μιλούν ε, για την αύξηση του αριθμού των αντιπροσωπιών ε, παγκοσμίως. Ε, πάντα με βάση βέβαια τους προώρους και τις προτεραιότητες. γιατί πραγματικά ε, αυτό που θα μας πούν είναι ότι αν θέλουμε ανοιχτές αυτές, να ανοίξουν αυτές οι αντιπροσωπείες θα πρέπει να βρούμε και τα μέσα να τις υποστηρίξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση και μετά να δούμε και τα οικονομικά μέσα που θα μας βοηθήσουν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λένε και οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ σχετικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Μπουριάν έχει δίκιο ότι πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε σε σχέση πάντοτε με τη στρατηγική για την Κεντρική Ασία. Είναι μια περιοχή που δεν θέλουμε να φύγει από τις προτεραιότητές μας και γι' αυτό καλωσορίζουμε την παρουσία του εδώ και τη συνεργασία του και στο μέλλον με το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλο. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπουριάννα, που είσαστε εδώ και ανταλλάσσετε απόψεις μαζί μας, αλλά και την κυρία Μανέσκου ευχαριστώ για την εξαιρετική και πολλή δουλειά που έχει αφιερώσει για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ενισχύσω λίγο αυτό που είπε μόλις ο συνάδελφος κύριος Χάουιτ. Έχουμε ανησυχίες εδώ που ε, δεν βελτιώνονται άμεσα ούτε από το γεγονός ότι τα γνωρίζουμε, ούτε από την έκθεση, ούτε από την παρουσίασή σας. Παρόλο που κατανοώ πλήρως ότι υπάρχει μια τάση η νέα ηγεσία του Τουρκμενιστάν να εμπλακεί πιο ε, πολύ με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω μια πιο στρατηγική ερώτηση. Είπατε ότι έχουμε λίγη δυνατότητα να κινήσουμε τα νήματα στο Τουρκμενιστάν. Μάλλον είμαι πεπισμένος ότι θα αυξηθεί αυτή η δυνατότητα χειρισμών μετά την έγκριση της συμφωνίας. Δεν θέλω να προκαταβάλω το μέλλον, όμως συνήθως με δύο τρόπους εξελίσσονται τα πράγματα. Όντως η συμφωνία δίνει ένα πλαίσιο για παράδειγμα για να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πούμε σε διάλογο με τις αρχές του Τουρκμενιστάν. Όμως οποιοδήποτε πλαίσιο ή αυτού του είδους απαιτεί και οι δύο πλευρές ε, να δρουν ενεργά για αυτό. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν μας εγγυάται κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι εκεί λοιπόν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτό το ζήτημα. Επίσης, ε, ρωτιέμαι αν η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για την κύρωση της συμφωνίας ε, από ότι να φτιάξει ένα πλαίσιο θεσμικό που να λειτουργεί. Οπότε όποιο σχόλιο και αν υποθεί από εμάς είναι καλοδεχούμενο. Γιατί ακόμα και εντός της Κεντρικής Ασίας αυτή η χώρα δεν είναι από τους ε, πρώτους ε, που υπερμάχονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Ασία. Επίσης, ε, στο άρθρο 7 μιλάμε για τις πολύ δειλές κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θεωρούμε ότι είναι ενθαρρυντικό σημάδι. Δεν θα μου άρεσε πολύ να βλέπω τέτοιες δηλώσεις ότι αυτές οι δηλές ε, μεταρρυθμίσεις είναι καλό σημάδι. Επίσης, το 10 λέει ε, για την συνεργασία με το Τουρκμεριστάν ως προς τη μεταχείριση των ε, κρατουμένων, αλλά στην ίδια παράγραφο παραδεχόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων, όχι τον καθεστώς, τον αριθμό τους. Υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω λοιπόν αν θα μπορούσα να υπερψηφίσω μια τέτοια σύσταση για κύρωση Παρόλο που πλήρως συμφωνώ και όλοι συμφωνούμε εδώ ότι πρέπει να εμπλακούμε στην περιοχή, περισσότερο δηλαδή στην Κεντρική Ασία και στο Τουρκμενιστάν. Όμως δεν ξέρω αν η κύρωση αυτή τη στιγμή είναι η βέλτιστη λύση για να πετύχουμε αυτή την εμπλοκή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μανέσκου που την προτίμασε. Πρόκειται για μια πλήρη έκθεση που ασχολείται με όλα τα κατάλληλα ζητήματα, ανθρώπινα δικαιώματα, περιφερειακή ασφάλεια, εμπόριο, συνεργασία, κράτος δικαίου. Νομίζω ότι αποτελεί πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση και παρά από τα σχόλια που έγιναν σε αυτή τη συζήτηση, εν τέλει θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια έκθεση που θα ψηφιστεί από την ευρεία πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Μπούριαν, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το έργο του στην περιοχή. Είναι σαφές σε όλους ότι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας θα πρέπει να είναι ενιαία. Και νομίζω ότι ο Πρεσβευτής Μπούριαν ακριβώς αυτό κάνει με τον ρόλο του. Αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων γίνεται καθώς θα συζητήσουμε την εφαρμογή της στρατηγικής για την Κεντρική Ασία στην Ολομέλεια. Εγώ, εκ μέρους της ομάδας μου, επαναλαμβάνω την έκκληση να έχουμε μία πλήρη αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν το συντομότερο. Κατανοώ τη λογική του, είπε ο κ. Βάσιριτς, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με ένα ρεαλιστικό τρόπο. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποια αναβολή θα κάνει καλό στη συνεργασία μας ε, με την περιοχή αυτή και άλλες περιοχές. Δεύτερον, πιστεύω ότι η θέση σε ισχύ τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία με το Τουρκμενιστάν θα βοηθήσει στο να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των σχέσεών μας. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε τα πράγματα αντικειμενικά, χωρί ε, να κάνουμε μεγαλοπίβολα σχέδια. Όμως και πάλι νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο και πιο πολύπλοκο διάλογο με τη χώρα. Δύο, τρία ερωτήματα στον κύριο Μπουρίαν και ίσως και στην κυρία Μανέσκου. Ξέρουμε ότι η κατάσταση στο Τουρκμενιστάν είναι ανησυχητική. Είναι ουσιαστικά ένα από τα πιο κλειστά καθεστώτα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Κεντρική Ασία. Όμως υπάρχουν κάποια σημάδια ότι υπάρχει κοινωνία των πολιτών είπατε. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, πόσο αποτελεσματικά το Τουρκμενιστάν ε, φυλά και διαχειρίζεται τα σύνορά του. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε ε, το project του Τουρκμενιστάν ε, για τα σύνορα και επίσης θα ήθελα να θέσω και μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Πώς αξιολογείται τη σημερινή κατάσταση της περιφερειακής συνεργασίας στην Κεντρική Ασία. Βλέπετε να υπάρχει μεγένθηση και αλληλοσύνδεση, τουλάχιστον ε, να, υπάρξει ένα περιβάλλον ασφαλείας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ κύριε Σμετίνη. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και τη συναδέλφο Μενέσκου για το έργο της. Ήταν μια δουλειά εις βάθος. Παραμένουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Εγώ κατανοώ την αξία της κύρωσης της συμφωνίας αυτής στο γεωπολιτικό επίπεδο και για να διατηρήσουμε και τις σχέσεις ε, με αυτή την ε, σημαντική χώρα. Επίσης είναι σημαντικό επειδή μιλάμε και για μια μουσουλμανική χώρα αποφασιστικής ε, σημασίας. Να μην είναι στη συνέχεια στην βορρά των εξτρεμιστών. Όμως το πρόβλημα που παραμένει επιτάπητος είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο ότι έχουμε μια αυταρχική χώρα χωρίς ελευθερίες και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν ε, νομίζω ότι τα βήματα που έχουν γίνει ήταν αποφασιστικά. Νομίζω ότι οι απαντήσεις ε, ήταν ανεπαρκείς. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και εγώ σκιώθηση εισηγητής για τη δική μου ομάδα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και κάποιες τροπολογίες που υπογραμμίζουν αυτή την πτυχή. Και αυτό γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Προς που για μας έχουν οικονομική σημασία που έχουν ε, τη δική τους ισχύ, τη δική τους δύναμη. Εμείς ε, μερικές φορές ε, είμαστε κάπως πιο ανεκτικοί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί. Και αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να είναι ολισθηρό έδαφος, γιατί ανάλογα με τις περιπτώσεις το κρίνουμε. Θα πρέπει, όπως και να έχει, να προσπαθούμε να διατηρούμε μια ισορροπία και να πράττουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρείται ένας κατάλληλος συνομιλητής. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και ελπίζω να μπορέσει να γίνει και αυτή η επικύρωση με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο. Euh, Σαφώς, ε, σύντομα κύριε Πρόεδρε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο προσεγγίσεις. μία αφορά τη δημοκρατία και η άλλη τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης. Τουλάχιστον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δύο προσεγγίσεις και αυτό συνιστά ήδη πρόοδο. Όχι μόνο δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα ή διπλωματία μάλλον από όχι ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, Πολλές φορές ε, εξαρτώνται τα πράγματα στο που βάζουμε τον κέρσορα, που βάζουμε το γνώμονα. Πρώτα είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ή πρώτα είναι τα οικονομικά ή στρατηγικά συμφέροντα. Και κάποιες φορές υπάρχει μια σύγχυση και κάποιοι ε, κινούνται με βάση τα δικά του συμφέροντα και όχι τα δικά μας συμφέροντα. Διαπιστώνω ότι συχνά έχουμε μια πολιτική μέτρων και δύο σταθμών στην έκθεση αυτή τουλάχιστον ε, υπάρχει τιμιότητα, αν θέλετε, του ότι το λέμε. Τη βάζουμε τον Κέρσορα, από τη μια στη Δημοκρατία και από την άλλη στα στρατηγικά συμφέροντα. Τώρα για να μιλήσω έτσι πιο γενικά, πιο σφαιρικά. Μετά από δύο χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύντομα, θα κλείσω τα δύο χρόνια, ε, διερωτώ με για την εξωτερική διάσταση της Ένωσης. Αν δούμε τον απολογισμό των διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων, εγώ πραγματικά διερωτώ με. Είναι χρήσιμο ή όχι τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι χρήσιμο ή δεν είναι χρήσιμη, είπατε εκπρόσωπος. Και οι πολιτικές μας συνολικά στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη συνεκτικότητας στις πολιτικές μας και τελικά ε, το πάνω χέρι το παίρνουν τα κράτη-μέλη. Να μιλήσω για την μεταναστευτική πολιτική, να δούμε τι έγινε με την Γερμανία που κάπως υπαγόρευσε αυτή την πολιτική και δεν είναι μεμονωμένη αυτή η περίπτωση. Το συναντάμε συχνά το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν πραγματικές στρατηγικές ή πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση αφενός μεταξύ της πολιτικής και των στρατηγικών συμφερόντων των κρατών μελών και αφετέρου μιας πιο σφαιρικής εικόνας, ενός πιο σφαιρικού οράματος των λαών της Ένωσης που ε, δυστυχώς διαπιστώνω και το λέω ξεκάθαρα και ισχύει για το Τουρκμενιστάν αλλά και σε πολλού άλλου τομείς ή περιοχές. Δεν μπορούμε να χαράξουμε ή να ορίσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Είτε πρόκειται για τον τομέα τη ενέργεια είτε τη μετανάστευση, αλλά μπορεί να πρόκειται τη διεύρυνση και για οποιοδήποτε άλλο τομέα. Πραγματικά λοιπόν μετά από δύο χρόνια διαρωτώ με για το κατά πόσον έχει νόημα να υπάρχει μια εξωτερική πολιτική. Εγώ είμαι Ευρωπαίος, παραμένω Ευρωπαίος, αλλά διαρωτώ με για τη χρησιμότητα ή μη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Das Κύριος Πέτερλε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουν και εγώ σε παρόμοια θέση πολλά χρόνια πριν, όταν είχα να αντιμετωπίσω το ίδιο θέμα, στο οποίο με διαδέχτηκε η συνάδελφος Ρεμόνα Μανέσκου. Η Και σκέφτομαι, ε, την... σε εύχομαι καλή επιτυχία. Η κατάσταση ως έχει λοιπόν μας ε, ε, υποδεικνύει να κάνουμε όχι αυτό που είναι το βέλτιστο, αλλά αυτό που είναι καλύτερο. Και αυτό που πρότεινε η συγγήτρια είναι καλύτερο από μια άλλη αναβολή. Και μέσα από αυτό θα βρούμε ένα εργαλείο για να επηρεάσουμε την κατάσταση. Στην έκθεση στην ουσία βλέπουμε ποιοι είναι οι τρόποι που θα εξελιχθεί η κατάσταση αν επιδεινωθεί. Για να ε, καταλήξω όσον αφορά στις αρχές που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι δεν είμαστε λιγότερο πραγματιστές από ότι ήμασταν σε άλλες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τολβοκλά. έχει το λόγο. Thank you, ο κύριος, ευχαριστώ. Είμαι επικεφαλής ε, του τμήματος για την Κεντρική Ασία από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Δεν θέλω να επαναλάβω ότι υπόθηκε εδώ. Από την εισηγήτρια ή από τον ειδικό εντεταλμένο. Απλώς ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία που σχετίζονται με την επιστολή που η Είπατε ότι εκπρόσωπο Μαντγκερίνη σας απέστειλε στα τέλη του περασμένου. έτους. Εκεί επανέλαβε τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί και από την προκατοχό τη για να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται δεόντως για την εφαρμογή των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του δημοκρατισμού στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Και επίση η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνεται απαραίτητο και είτε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είτε στην ε, πλαίσιο της αντιπροσωπείας. Και σήμερα ε, ο διόλογος γίνεται και σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων έχουμε ένα τμήμα τη ετήσια έκθεση για το Τουρκμενιστάν. Αλλά επίση είμαστε έτοιμοι να έχουμε ανταλλαγή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επόμενη στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το Τουρκμενιστάν που προετοιμάζεται φέτο από τον επικεφαλή τη αποστολή στο Ασκαμπάτ. Και θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, κατόπιν τη επίσκεψη των τριών μελών τη επιτροπή σα ε, στο Σκαμπάτ ε, το Μάιο και για να συζητήσουμε ρεαλιστικά σημεία για πρόοδο για τα επομενα τρία 3-5 έτη. Οι στρατηγικές των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δημόσια έγγραφα, αλλά διαβουλεύσεις με τους βουλευτές θα μπορούσαν να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας. Εμείς θεωρούμε ότι η PCA δεν είναι σκοπός, αλλά ένα εργαλείο για καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να πετύχουμε αυτούς τους κοινού σκοπούς που έχουμε όλοι, δηλαδή μεγαλύτερος εκδημοκρατισμός και πιο ανοιχτός χαρακτήρας στο Τουρκμενιστάν. Αυτά θα επιτευχθούν αν έχουμε έναν ισχυρό και συνεχή διάλογο με αυτή τη χώρα, φυσικά και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Godātie kolēģi, um, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και πρέπει να σας πω ότι πέρυσι για πρώτη φορά η επίσημη αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωκοινοβουλίου ήρθε για συνομιλίες μαζί μας ε, με ευρωβουλευτές. Και ένα από τα ζητήματα, τα βασικά ζητήματα που συζητήσαμε ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις συζητήσεις μας ε, με τις χώρες ε, από τη Ανατολή εστιάζουμε στα εργαλεία τα οποία έχουμε και στις βάσεις που δεν έχουμε πει. Το Σεπτέμβριο Θα έχουμε μία αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν για να αρχίσει μια πολύ καλή πρακτική. Φυσικά, πολύ πριν ε, ε είπανε ότι συμφωνούν πως ε, αυτή η συμφωνία πρέπει να κυρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία ε, θετικά διότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο αυτή η συμφωνία, θα πάρουμε πράγματα από αυτήν. Όμως θεωρώ ότι γενικά ε, καλό είναι να κάνουμε κάτι παρά να μην κάνουμε τίποτα και να επικρίνουμε. Γι' αυτό ζητώ από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή την έκθεση για να μπορέσει πραγματικά να πραγματοθεί αυτή η κύρωση ε, ε, πέρασε πολύ καιρό, ε, πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Στην Κεντρική Ασία, αν θέλουμε να παίξουμε έναν ρόλο, πρέπει να είμαστε προμηθείς. Δεν μπορούμε απλώς να βάζουμε πράγματα στο σιρτάρι και να περιμένουμε τους άλλους ε, να δράσουν πρώτοι. Θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα είναι οι πιο έξυπνοι, οι πιο δυνατοί, οι πιο ε, πεπειραμένοι πρέπει να δείξουμε πώς πρέπει κανείς ε, να φτιάξει μια δημοκρατική κοινωνία, πώς να εκπροσωπεί τις δημοκρατικές αξίες και γι' αυτό θέλω να υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί θεωρώ ότι η έκθεση μας προετοιμάζει πολύ καλά για την τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το 2011 Ήδη συζητήσαμε το θέμα αυτό και την αρισιμότητα και έχει τώρα λήξει η νομική βάση. Ε, αυτό λοιπόν που υπογράψαμε δεν έχει πάει στην Ολομέλεια. Θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να συζητούνται στο Κοινοβούλιο και σε αυτό το διάλογο να συμμετέχει και η κοινωνία των ε, πολιτών και γι' αυτό ε, στείλαμε μια επιστολή τον Σεπτέμβριο στην κυρία Μοργκερίνη που ε, και αυτή μας απάντησε ότι ε, θα υπάρχει μια συνομιλία για να υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις έτσι ώστε Ε, η δεύτερη ανάγνωση του έκθεσης ε, να γίνει στις 14 Μαΐου, δηλαδή μια εβδομάδα μετά το ταξίδι στο Τουρκμενιστάν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί στην ΕΙΑΔ και να συζητήσουμε κι εμείς ε, μεταξύ μας, να δούμε πώς θα πάρουμε τη δική μας απόφαση σχετικά με αυτήν την διαδικασία Όταν γυρίσουν οι συνάδελφοι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, που θα, μας, ε, ε, θα γίνει και η σχετική ενημέρωση και θα μπορεί να πάει στην Ολομέλεια η έκθεση έτσι ώστε να ξεκινήσει η αντιπροσωπεία για να είμαστε σε καλύτερη θέση να παρακολουθήσουμε αυτό το διάλογο και να επηρεάσουμε αυτό το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ Λοιπόν, ε, πριν φτάσουμε σε οποιαδήποτε απόφαση, μετά τις ε, συζητήσεις το Μάιο, να ακούσουμε την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο, κυρία Μανέσκου. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους όσους όλους όσοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους, αλλά και τις ανησυχίες τους σε σχέση με την κατάσταση στο Τουρκουμενιστάν και την υποστήριξή τους προς τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Πιστεύω ότι θα είμαστε επικοδομητικοί μετά από 16 χρόνια αναβολών και ουσιαστικά καμία ουσιαστική ε, αλλαγή στο ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε τώρα ότι έχουμε πια έναν εταίρο, έναν συνομιλητή που φαίνεται να είναι πιο ανοιχτός και πιο πρόθυμος ε, για συνεργασία μαζί μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη και να το θεωρήσουμε θετικό σημάδι, να το ενθαρρύνουμε. Για να ενθαρρύνουμε το Τουρκμενιστάν να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε. Ρώτησε ο πρόεδρος αν η επιστολή της ΕΠΑΤΣ εκπροσώπου ήταν ικανοποιητική. Ναι, ήταν. Ακριβώς αυτό είχαμε ζητήσει. Έναν μηχανισμό, ένα εργαλείο παρακολούθησης και συμμετοχής μαζί με την Κομισιόν στην όλη αυτή διαδικασία. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να επωφεληθούμε της ύπαρξης αυτού του νέου εργαλείου. να εμπλακούμε λοιπόν στην όλη διαδικασία μαζί με την Κομισιόν πριν την αποστολή. Υπάρχει στις 17 Μαΐου και ο διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε βεβαίως να ζητήσουμε από την ΕΙΕΔ να μας στείλει την έκβαση αυτού του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να είμαστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει και για την πρόοδο που συντελείται στο Τουρκμενιστάν. Νομίζω ότι όλους μας απασχολούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι θέλουμε να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Έχουμε ένα κατάλογο, τον λάβαμε από τις αρχές. Αλλά όλα αυτά είναι λόγοι παραπάνω για να είμαστε παρόντες και να πιέζουμε τις αρχές του Τουρκμενιστάν. Να κάνουν περισσότερα και να τα κάνουν και πιο γρήγορα, γιατί φυσικά και είναι βραδείς. Δεν περιμένουμε ε, μια νυχτή να έχουμε μια καταπληκτική δημοκρατία στη χώρα. Μπορούμε όμως να τους υποστηρίξουμε στο δρόμο να γίνουν μια δημοκρατική χώρα. Νομίζω ότι η συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Και τουλάχιστον ε, για τις αρχές του Τουρκμενιστάν συνιστά υποχρέωση, δέσμευση να συνεχίσουν το διάλογό τους, το διάλογό τους μαζί μας και να σεβαστούν τις υποχρεωτικές διατάξεις της συμφωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν όλες τις, τις διατάξεις, να, να σεβαστούν όλες τις διατάξεις της συμφωνίας. Και εμείς θα τα παρακολουθούμε αυτά με τους εμπειρογνώμονες μας. Φυσικά είναι, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα συναντήσεων, διαλόγου στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν το είχαμε προηγουμένως. Άρα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να το θεωρήσουμε ένα εργαλείο. Γιατί πολλοί συνάδελφοι είπαν και ρώτησαν τι παραπάνω προσφέρει αυτή η συμφωνία. Θα είμαστε εκεί λοιπόν και θα τους παρέχουμε καθοδήγηση. Το είπαν αρκετοί συνάδελφοι. Θα τους παρέχουμε καθοδήγηση έχοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα σημεία αναφοράς, όλα τα benchmarks που συνοδεύουν τη συμφωνία στο ψήφισμα είναι σημαντική, σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι σημαντικό το ψήφισμα αυτό, μαζί με το ψήφισμα για την ε, επικύρωση, γιατί στο ψήφισμα αυτό αναφέρουμε ξεκάθαρα τις προσδοκίες μας, ε, τις ε, απαιτήσει μας και φυσικά εκφράζουμε και την στήριξή μας προς τις αρχές του Τουρκμενιστάν, από τις οποίες ζητούμε να προχωρήσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και είναι αυτό κάτι πιο θετικό και πιο επικοδομητικό από τις συνεχείς αναβολές ή το να αφήνουμε μόνο το, το Τουρκμενιστάν να λύσει τα προβλήματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δούμε την επόμενη φορά. 23 είναι η προθεσμία για την ε, εξέταση των τροπολογιών. 18 Απριλίου λίγη προθεσμία για την κατάρτιση τροπολογιών και πάμε στην Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή. Ο κύριος Οστρεβίτσιους που τα ελέγχει όλα εκεί. Ευχαριστώ αγαπητοί σκιώδεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκ μέρους του εισηγητή του Χαβιενάρτ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του σε αυτή την συνεδρίαση και να παρουσιάσω εν συντομία τις κυρίες ιδέες της έκθεσης για την πρόταση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η πρόταση αυτή προσπαθεί να προωθήσει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες της σημερινής Frontex και θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα σταδιακό πρώτο βήμα προς μια πλήρως διαφανή και ολοκληρωμένη συνοριοφυλακή και εκτοφυλακή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει επιχειρησιακή αυτονομία και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεισφορά και συνεργασία των κρατών μελών ε, είναι ζωτικό θέμα στην έκθεση αυτή προκειμένου να διασφαλίσουμε πλήρη αποτελεσματικότητα για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει στα εξωτερικά σύνορα. Έτσι θα πρέπει να αναμένουμε σαφή πολιτική δέσμευση από τα κράτη-μέλη στο πρακτικό τομέα. Όπως ε, δηλώνεται, στην έκθεση ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω για να ξεκαθαρίσουμε την έννοια των μερισμένων ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συνοριοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούν να υπάρχουν ασάφειες στον τομέα αυτό. Μία σειρά τροπολογιών έχουν ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, καθώς και να καταστήσουν σαφές ότι οι καλές σχέσεις με τις τρίτες χώρες είναι απαραίτητοι. Μεταξύ άλλων τροπολογιών που προτείνονται από αυτή την Επιτροπή, ε, είναι και οι τροπολογίες για την αποσαφήνιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβαίνει σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων και αξιολογήσεις ε, προκειμένου να γίνουν σεβαστές όλες οι πτυχές του κανονισμού. Τέλος, ο συνάδελφος ε, ε, ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για το ότι ακολουθείτε εδώ μία διαδικασία ταχύτατη ε, καθώς είμαστε μεσούσεις της προσφυγικής κρίσης. Ε, ε, βέβαια, καλωσορίζει τις προσπάθειες να έχουμε περαιτέρω προθεσμία και για την κατάθεση αλλά και για την έγκριση της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας εκ μέρους του. Και αναμένω σχόλια ή ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο γιατί θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στη συνεδρίαση του Μαΐου. Νομίζω έχουμε μια συνεδρίαση και με τον Πρωθυπουργό της Βοσνίας. Και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε τροπολογίες. Concerns στις 14 Απριλίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Έτσι λοιπόν, στις 12 Μαΐου στην έκτακτη συνεδρίαση μπορούμε να ψηφίσουμε. Και η ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου. Είναι καλύτερη λοιπόν η κατάσταση τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτή είναι η πρότασή μου λοιπόν έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων πριν να ψηφίσουμε στις 12 Μαΐου. Ποιος θέλει το λόγο, κύριο Στεκίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Να σας πω ότι υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής. Θεωρώ ότι αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα εξωτερικά μας σύνορα. Με λίγα λόγια να πω ότι η Frontex ε, ως έχει δεν είναι σε θέση να αντιδράσει αποτελεσματικά στις μεταναστευτικές ροές ε, με τον τρόπο που έχουν εξελιχθεί φέτος στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να υποστηρίξουμε μια νέα λύση. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση μιας επιταχυμένης διαδικασίας και χαίρομαι και για τις σύντομες προθεσμίες που έχουμε για την κατάθεση των τροπολογιών. Όσον αφορά τώρα στην ε, αρμοδιότητα της άλλης επιτροπής χαιρετίζω που το σχέδιο της πρότασης ε, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της συνεργειακής και των τρίτων χωρών. Μπορούμε ας πούμε να στείλουμε ε, liaison ε, officers, δηλαδή αξιωματικούς συνδέσμους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες το πεδίο της συνδρομής ε, που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέχει σε τρίτες χώρες όσον αφορά στην προστασία και την επιστροφή των μεταναστών πρέπει να είναι το ευρύτερο δυνατό. Αυτό θα πρέπει να μας βοηθήσει να διευκολύνουμε την συνεργασία με τις τρίτες ε, χώρες και με τις γραπτές ε, επιχειρήσεις. Ε, γι' αυτό λοιπόν αδειμονώ ε, να συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ για την... Ευχαριστούμε τον κύριο Αστραβίσιους. Να σας πω ε, ότι η δουλειά του εισηγητή και των σκιωδών είναι πολύ καλή και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει άλλη συνεδρίαση μέχρι τις 12 Μαΐου, οπότε θα μπορούμε να έχουμε διαλευκάνει όλα τα ζητήματα. Ο κύριος Πίτσουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του εισηγητή για την πολύ καλή και συνοπτική άποψη που εκπροσωπεί τις απόψεις του και του Συμβουλίου. Ε, να πω ότι συμφωνώ ότι ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες σε, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια πιο φιλόδοξη λύση. Αν θέλουμε να έχουμε ε, κοινή ευθύνη, όπως λέγεται, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την προηγούμενη κατάσταση με τα σύνορα. Ε, όλα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή, με την εκτέλεση. Όταν έχουμε λοιπόν μια πρόταση για μια κοινή υπηρεσία, έναν κοινό οργανισμό για τα εξωτερικά σύνορα επί, ε, επί της ξηράς και επί της θάλασσας, πρέπει να την υποστηρίξουμε. Όμως πρέπει τα στοιχεία που δεν είναι διευκρινισμένα να τα διευκρινίσουμε, ας πούμε, να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τις ευθύνες του οργανισμού και ποιοι θα είναι αυτοί που θα εργάζονται εκεί, πόσοι θα είναι, πόσο θα πληρώνονται. Μετά, η επικουρικότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, θέμα που θα χρησιμοποιηθεί και στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Ε, η δομή, οι αρμοδιότητες είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενδεχομένως. Ε, θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να το συζητήσουμε μέχρι τέλος γιατί είναι πολύ σημαντικό για πολλά κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να ορίσουμε και τον χώρο που θα ορίζεται στο άρθρο 12.3 μιλάμε για το vulnerability, την τροτότητα. Εκεί ε, ε, στην ουσία λαμβάνεται υπόψη ο χώρος Σέγγεν, όμως το άρθρο 1.1 ε, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση που απειλείται ο χώρος του Σέγγεν μπορεί η Κομισιόν να πάρει μέτρα τα οποία θα την βοηθήσουν να προστατεύσει αυτόν τον χώρο. Νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που πιστεύει πως αυτό το νέο ολοκληρωμένο σύστημα για τα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να προστατεύει όλους την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο αυτούς που εντάσσονται στο ΣΕΝΚΕΤ, όλους την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το σύστημα που έχουμε ως τώρα είναι κάτι που ε, δεν είναι ικανοποιημένο ο εισηγητής με αυτό και θα επαναληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία και πρέπει να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε συνάδελφοι, είναι περιττό να επισημάνω το πόσο σοβαρό είναι ο κανονισμό που συζητάμε σήμερα. Επίση, με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νάρτ για την διεξοδική προσέγγιση που έχει κάνει και την ανταπόκριση που έδειξε στο αίτημά μου για περισσότερο χρόνο, ώστε να ανταποκριθούμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα ε, σε αυτόν τον κανονισμό. Γνωρίζετε την αντίθεση της πολιτικής μου ομάδας όσον αφορά στην ίδρυση και στη λειτουργία της Frontex, όμως παρά τις πολιτικές ανησυχίες μας και τις επιφυλάξεις για τον κανονισμό, προσωπικά είμαι διατεθειμένη να συνεισφέρω όσο μπορώ ώστε να καταλήξουμε και αν είναι δυνατόν σε κοινέ θέσεις και σε προτάσεις με δεδομένα τα πολύ σοβαρά και λεπτά ζητήματα στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός και για να ξεπεράσουμε διαφορετικές πολιτικές οπτικές, πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο και με γνώμονα τα όσα προστάζουν οι διεθνείς ε, συνθήκες. Εκτιμώ ότι είναι το ελάχιστο πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε, με δεδομένο ότι η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση στην Ευρώπη, και ενώ τα κλειστά σύνορα, τη συμφωνία με την Τουρκία η οποία παραβιάζει συνεχώ τη ε, διεθνή νομιμότητα, υψηλή τόνη αντιπαράθεση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και άλλα, αλλά και γεγονότα που επιβεβαιώνουν ανησυχίε και φόβου, παραδείγματο χάρη οι φυλακίσει των επαναπροωθέντων στην ε, Τουρκία προσφύγων, αλλά και τα περιστατικά βία κατά αυτών, μας αφαιρούν νομίζω οποιοδήποτε δικαίωμα στο να ολιγορήσουμε. Είναι πασιφανές ότι αυτός ο κανονισμός δεν έρχεται να αντιμετωπίσει στατικά ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αλλά ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου θα διωγγώνεται και θα οξύνεται με την πάροδο του χρόνου και άρα έχουμε ευθύνη και για τη μελλοντική του λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τελειώνοντας, θα αναφερθώ σε τέσσερα-πέντε θέματα, στα οποία και θα εστιάσω τις παρεμβάσεις και τις τροπολογίες μας πρώτον στην ενεργή συμμετοχή και τον έλεγχο που θα πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο στα ερετά όργανα του οργανισμού και που θα πρέπει να είναι ενισχυμένος και διασφαλισμένος, στην δικαιοδοσία του σώματος αλλά και το φάσμα των επιχειρησιακών παρεμβάσεων που θα πρέπει να είναι απόλυτα διευκρινισμένο έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση να μην έρθει σε σύγκρουση με τις υπάρχουσες συνθήκες, Επίσης το γεγονός ότι στη σημερινή συγκαιρία οι πόροι χρηματοδότησης του οργανισμού και η διαχείρισή τους οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως την αναλογικότητα και την διαφάνεια και να επισημάνω την κάθετη αντίθεσή μου στη διαφαινόμενη πρόθεση να ελέγχει ο οργανισμός προγράμματα όπως είναι το Horizon 2020, τα οποία ήδη τρέχουν αλλά και μελλοντικά με ιδιαίτερα υψηλούς προϋπολογισμούς. Και κλείνοντας, τέλος, να επισημάνω την ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί σε θέματα που αφορούν στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία των εθνικών κρατών μελών και να εκφράσω τον ιδιαίτερο προβληματισμό μου όταν σε ένα τέτοιο κέρια σημασία κανονισμό δεν περιγράφονται με σαφήνεια, κύριοι συνάδελφοι, ποια σύνορα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σαν εξωτερικά τη σύνορα. Και θέλω να συγχαρώ ξανά τον κύριο Νάρτ που τα επεσήμανε με την τροπολογία του που είναι και ακριβέστατη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαλέρο. Eh, eh, <clears throat> Ευχαριστώ. Αυτό το ζήτημα πραγματικά με χαροποιεί, διότι έχουμε κάποιες μέρες ε, μέχρι να καταθέσουμε τις τροπολογίες, καθώς είναι ήδη αργά και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μας έκανε την παρουσίαση αυτή. Το πρόβλημα είναι το κείμενο του κανονισμού. Αν ε, διαβάσει κανείς την αιτιολόγηση θα δει ότι αυτά που βρίσκονται στα άρθρα ε, αντιφάσκουν με αυτά που λέει η αιτιολόγηση. Αυτό που έχει να κάνει με το σκοπό ή τον προϋπολογισμό. Δεν θα πρέπει να είναι πιο μεγάλος από ό,τι στο παρελθόν, αλλά μετά γίνεται αναφορά στις ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών και ε, ως στόχος αναφέρεται ότι θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση της μετανάστευσης, όχι οι ανθρώπινες ζωές. Αυτές οι αντιφάσεις, ε, ειδικά ως προς το σκοπό, είναι κάτι που θέλω να, να μπορέσω να διορθώσω με τις τροπολογίες μου. Να υπάρχει η διάσωση ανθρωπίνων ζωών στο σκοπό. Επίσης, να ε, σταματήσουν οι διάφορες αντιφάσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων άρθρων. Κάπου λέει, για παράδειγμα, ότι δεν όταν δεν πρέπει να αμφισβητούμε τον τρολόγο για τον οποίο θέλουμε να επαναπροωθήσουμε κάποιον. Ε, όμως ε, ε, κάπου αλλού αναφέρεται ότι πρέπει να δούμε πώς είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διάφορες χώρες όπου στέλνονται οι άνθρωποι. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Επίσης αναφέρεται ότι πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα να τηρούνται. Είναι σημεία λοιπόν που φάσκουν και αντιφάσκουν και θα πρέπει να τα διορθώσουμε. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αυτά που κάνουμε πρέπει να είναι σύμφωνα με το δημόσιο και ε, με το διεθνές δίκαιο. Και πολύ σπάνια ο Γενικός Διευθυντής έχει έναν τόσο ισχυρό ρόλο και μια τόσο ισχυρή εντολή ακόμα και κατά της θέλησης των ε, κρατών μελών να μπορεί να παίρνει μέτρα. Αυτά είναι θέματα που θα αμφισβητηθούν. Ένας γενικός διευθυντής θα πρέπει τουλάχιστον να ε, μπορεί να στρέφεται στο Προεδρείο και εκεί να μπορεί να συζητά τις θέσεις των κρατών μελών. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να καταθέσω πολλές τροπολογίες και αυτές ε, στην ουσία θα έχουν να κάνουν με τη διάσωση ανθρωπίνων ζώων. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι γεγονός ότι οι ξαφνικές, ανεξέλεγκτες και μεγάλες ροές των παρανόμων μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα κάτι για το οποίο η Τουρκία δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποτρέψει, μας υποχρεώνουν να πάρουμε βεβαιασμένες αποφάσεις οι οποίες δεν πρόκειται κατά την άποψή μου να επιλύσουν το πρόβλημα. Απλά θα πάρουμε μία ασπιρίνη για να αντιμετωπίσουμε μία σοβαρή ασθένεια που θέλει ισχυρό αντιβιωτικό. Επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την προσέγγιση. η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων κάποιου κράτους. Τα κράτη πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο και την ασφάλεια των συνόρων τους και όταν αυτά είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, η ευθύνη των κρατών αυξάνεται. Όταν το κράτος, τα σύνορα του οποίου είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διαπιστώσει πως χρειάζεται κάποια βοήθεια αυτή η βοήθεια θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι επιβοηθητικός και όχι πρωταρχικός. Δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε ένα ακόμη αναποτελεσματικό οργανισμό ο οποίος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι η κατά επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Η εμπειρία του Frontex πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Δεν εξυπηρετεί τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων η δημιουργία μιας υπηρεσίας καταγραφής. Εκείνο που απαιτείται είναι η δυνατότητα αποτροπής της εισόδου παρανόμων μεταναστών στο έδαφος ενός κράτους και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό όμως, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί να το επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή. Αυτό προκύπτει και από την οργάνωση και την αποστολή αυτού του οργανισμού. Ακόμη περισσότερο είναι απαράδεκτη η πρόβλεψη του άρθρου 18 του κανονισμού που αναφέρεται στη δημιουργία της συνοριοφυλακής ακτοφυλακής να μπορεί δηλαδή να επεμβαίνει αυτή αυτοβούλος κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής ακόμη και όταν το ενδιαφερόμενο κράτος δεν συνενεί. Πέραν του ότι καταργείται η κυριαρχία του κράτους και αυτό είναι απαράδεκτο δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Πολύ απλά διότι αυτή η συνοριοφυλακή δεν έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει, όπως είπα και προηγουμένως, την παράνομη είσοδο ατόμων σε ένα κράτος. Εδώ το ΝΑΤΟ το οποίο είναι αμυντικός οργανισμός, άρα έχει πολύ καλύτερη οργάνωση, έχει αποτύχει παταγωδός στο Αιγαίο. Και μη σας φαίνεται παράξενο αυτό, δεν έχει κατορθώσει να εμποδίσει την ε, ροή των παρανόμων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν κατά μείζωνα λόγο δεν μπορεί να επιτύχει αυτό αυτός ο οργανισμός που θέλουμε να δημιουργήσουμε, συνοριοφυλακής, αγροφυλακής. Συμπερασματικά μπορώ να πω ότι ένα πρόβλημα δεν επιλύεται ούτε με ιδεολειψίες, ούτε με φαντασιώσεις, ούτε με προσπάθειες να προωθήσουμε πολιτικές σκοπιμότητες. Επιλύεται με αντικειμενική ανάλυση του προβλήματος και επιλογή μέτρων πραγματιστικών και εφαρμόσιμων. Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έχω κάνει πολλές προτάσεις οι ανθρωπολογίες και θα το παρακολουθώ στενά, οπότε θα με ακούσετε και άλλη φορά να παρεμβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ. Ο εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων που όλοι ακούσαμε. Φυσικά και θα διαβιβάσω τις σημειώσεις μου ε, στον ε, συνάδελφο Νάρτ. Δεν έχει μείνει πολύ χρόνος, τρεις μέρες. Ε, φαντάζομαι θα έχουμε και άλλες τροπολογίες. Θα έχουμε και μια ακόμη πιο αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων. Όλα αυτά πιστεύω και ελπίζω ότι θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μας να έχουμε ένα κείμενο <clears throat> το οποίο θα μπορεί να το υποστηρίξουν περισσότεροι. Το βέλτιστο δυνατό δηλαδή. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα από ό,τι βλέπω. Οπότε σας εύχομαι καλό βράδυ. Τελειώνουμε εδώ.